Okay, so dear colleagues, I think we can start the meeting. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir... Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε τη σημερινή μας συνεδρίαση. Και περνάμε κατευθείαν στην ημερήσια διάταξη. Σημείο 1. Έγκριση της μερικής διάταξης. Την ε, εγκρίνουμε αν δεν υπάρχουν ενστάσεις. Περνάμε στις ανακοινώσεις του Προέδρου. Ε, είναι web streamed η συνεδρίασή μας. Σε 20 γλώσσες έχουμε διερμηνία. Η επόμενη συνεδρία προβλέπεται για τις 6 Ιανουαρίου του 2020. Δεν θα λάβει χώρα όμως τελικά, γιατί δεν υπάρχει επίγουσα ανάγκη. Και επίσης να σας πω ότι σήμερα το απόγευμα μετά τη συνεδρίαση θα έχουμε κοκτέιλ αμέσως μετά τη συνεδρίαση. Ένα άτυπο για το τέλος του έτους, ώστε να έρθουμε σε επαφή μεταξύ μας. Περνάμε στο πρώτο ε, θέμα. Απαλλαγή 2018, Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα δώσω το λόγο στον ε, εισηγητή, στον ε, κύριο Κόβατς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος, γιατί έχω να κάνω μία ακόμα παρουσίαση μέσω μετά από αυτήν και θα μιλήσω στην μετρική μου γλώσσα στα Ουγγρικά. Προσπάθησα να κρατήσω μια ισορροπία στην διατύπωση και να ε, τονίσω τα πιο σημαντικά σημεία. Είχα όμως ε, να αντιμετωπίσω και κάποια συγκεκριμένα πράγματα, όπως την έκταση, το μέγεθος του εγγράφου. Αυτά όμως που δεν μπόρεσα να διατυπώσω, για αυτά που δεν μπόρεσα να διατυπώσω, θα σας θα υποβάλω ε, τροπολογίες και περιμένω και τις δικές μέχρι, τις, μέχρι την 6 Δεκεμβρίου. Περί τίνος πρόκειται σε αυτή την πρόταση, λοιπόν. Ε, επιδοκιμάζουμε τα πόρισματα του ελληνικτικού συνεδρίου ότι όλα ε, έγιναν σωστά και το ποσοστό των λαθών δεν είναι πάνω από το 2,4%. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι τηρήθηκαν οι προδιαγραφές για την ευζοία των ζώων. Έχω ανησυχίες και τις εκφράζω. Ότι έχουν γίνει φαρπαγές γης από ολιγάρχες και κάνω λόγο και για την, ε, τον κίνδυνο της επαθηνικοποίησης της ε, κοινή ε, γεωργικής πολιτικής και επίσης κάνουμε λόγο για μια πράσινη κοινή γεωργική πολιτική. Παράλληλα τονίζω ότι είναι εξίσου σημαντική η υποστήριξη των νέων γεωργών και αυτό μπορεί να γίνει με την απλούστευση των κανόνων και με την διευκόλυνση στο διοικητικό κομμάτι. Έκανα αναφορά στις τροπολογίες. Θα ήθελα να παρακαλέσω την Επιτροπή όσον αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη να αυξήσει το ποσοστό εκτέλεσης, το ποσοστό απορρόφησης συγκεκριμένων το ε, αυξήσει. Επίσης, πολύ σημαντική είναι η ψηφιοποίηση της ε, γεωργίας. Τα smart farms και τα smart villages και τα προγράμματα τα σχετικά ε, ήδη τρέχουν και θα πρέπει να βελτιστοποιηθούν. Και τέλος, θα ήθελα ε, να υπάρχει δίκαιη και ισότιμη κατανομή μεταξύ κρατών μελών. Είναι ένα σύντομο ε, κείμενο σε γενικές γραμμές. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Yeah, Σας ευχαριστώ, κύριε εισηγητή. Περνάμε στους σκιώδεις εισηγητής από το ΕΛΚ, ο συνάδελφος Ντόρφμαν. Ευχαριστώ πολύ. Θα πω εν συντομία Να ευχαριστήσω αρχικά τον εισηγητή για την επικοδομητική συνεργασία στην σύνταξη αυτής της ε, γνωμοδότησης. Συμφωνώ με την ε, άποψή του. Δεν έχουμε αντιρρήσεις ως ΕΛΚ με αυτή την πρότασή του. Όσον αφορά την ε, απαλλαγή, τις απαλλαγές, ε, θα μπορούσε σε αυτό το σημείο να βελτιωθεί κάπως το έγγραφο, αλλά κατά τα άλλα είμαστε εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, συνάδελφος Κρίστενσεν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή μας για το σχέδιο γνωμοδότησης που υπέβαλε. Θα ήθελα να τονίσω ότι το ολοκληρωμένο ε, σύστημα ελέγχου είναι απαραίτητο για τη μείωση του αριθμού των σφαλμάτων στο σύστημα και στο μέλλον θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ε, στην εφαρμογή της ΚΑΠ μετά το 2020. Γι' αυτό θα πρέπει να στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διαπραγμάτευση συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών που θα πρέπει όμως να είναι φιλόδοξες, ε, δίκες και ισορροπημένες. Και επίσης θα πάνε απέναντι στις ε, χώρες εντάρρους με τις οποίες διαπραγματευόμαστε θα πρέπει να απαιτήσουμε τη συμπερίληψη ενός χάρτη βιωσιμότητας στις εμπορικές συμφωνίες μας. Επίση θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τι ενισχύσει τη γεωργία και να υπάρχει διαφάνεια και προ την ιδιοκτησία τη γη. Στη Δανία κάθε ε, χρόνο έχουμε έκθεση για το ύψος των ενισχύσεων που λαμβάνει ο κάθε γεωργός και ενημέρωση για την κυριότητα των ε, γεών του. Έτσι υπάρχει διαφάνεια. Θέλουμε καλύτερους δείκτες βιωσιμότητας. Και επίσης καλύτερη χρησιμότητα των σφαλμάτων στην ΚΑΠ μετά το 2020. Θα πρέπει και η ΚΑΠ να συμβάλλει στο μετριασμό των κλιματικών αλλαγών σίγουρα. Και το κρίσιμο εδώ είναι να αναπτύξουμε περισσότερες φιλοπεριβαλλοντικές τεχνολογίες και μάλιστα ως ύψητη προτεραιότητά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και ο συνάδελφος Χόισλινγκ. Ευχαριστώ. Δεν θα υποβάλω πολλές τροπολογίες, αλλά θα μιλήσω για μια έκθεση, μια, ένα άρθρο New York Times όσον αφορά τις κατηγορίες για την ε, διαφθορά στις ευρωπαϊκές χώρες είναι κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε γιατί αποτελεί πλήγμα για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το που διοχετεύονται τα ε, κονδύλια. Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε θα έχουμε πρόβλημα ε, απώλειας της αξιοπιστίας στην κοινή πολιτική. Θα πρέπει να ε, δούμε και τους νέους στόχους της Επιτροπής ε, και θα υποβάλουμε και για αυτούς ε, κάποιες σχετικέ τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Κούτσμιεκ. Δεν πρόκειται να καταθέσω καμία τροπολογία στο σχέδιο γνωμοδότησης ούτε από το, την πολιτική μου ομάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από τις υπόλοιπες ομάδες δεν ε, βλέπω κάποιους ε, εισηγητές. Θα ήθελε κάποιος να πάρει το λόγο. Από τις άλλες πολιτικές ομάδες ή κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Όχι. Θα δώσω και πάλι λοιπόν το λόγο στον ε, εισηγητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βλέπω την υποστήριξή σας. Ιδεολογικά μπορεί να διαφέρουμε σε κάποια πράγματα, αλλά εδώ υπάρχει, εδώ συμφωνούμε. Ο στόχος μου όταν συνέταξα αυτή την πρόταση ήταν να, υπάρξει, να υπάρχει ισορροπία και βλέπω ότι κάθε ομάδα βρήκε κάτι χρήσιμο και αυτό που θέλουμε όλοι είναι την βελτίωση της κοινή αγροτικής πολιτικής, οπότε έχουμε ένα κοινό στόχο. Ευχαριστώ. Ξέχασα να δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Παρακαλώ. Thank you, Chair. Uh, my name is Christina Ευχαριστώ. Ονομάζομαι Κριστίνα Μπόργμαν και είμαι Διευθύντρια για την Ασφάλεια και τον Έλεγχο στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Σε ό,τι αφορά την τη δήλωση αξιοπιστίας, νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο επίπεδο ε, εξασφάλισης ε, ε, στην κοινή πολιτική, κάτι που φαίνεται από το χαμηλό ποσοστό σφαλμάτων. Και μάλιστα και το δικαστήριο είπε ότι οι άμεσες ενισχύσεις ε, από το γεωρικό Ταμείο δεν συνιστούν δαπάνες αγοράς. Οπότε ε, και, όπως λέει και το Ελεκτικό Συνέδριο, δεν υπάρχει για το γεωρικό Ταμείο ουσιαστικό σφάλμα. Και σας ευχαριστώ που αναγνωρίζετε την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διόρθωση. Ο εισηγητής ε, χαρακτήρισε ιδιαίτερα μακροσκελές το έγγραφο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε και την απάντηση όμως επισυνημένη στην έκθεση. Και όταν βλέπετε για το πλαίσιο επιδόσεων και ζητάτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να το εγκρίνει, εμεί έχουμε ήδη δεχτεί τη σχετική σύσταση. Και στην απάντησή μα επισημαίνουμε ότι το όλο σύστημα επιδόσεων μετά το 2020 βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση με του ε, συνομοθέτες, δηλαδή και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό ισχύει και για τον οριζόντιο κανονισμό και το κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια. Έχουμε, έχουμε ήδη δηλαδή διαβιβάσει την απάντησή μας. Επίσης, για την ΚΑΠ μετά το 2020. Θα ήθελα να πω το εξή. Ζητάτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποτρέψει την επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ. Εμείς θεωρούμε ότι η πρότασή μας για μετά το 2020 εξασφαλίζει ένα πεδίο ίσων συνθηκών ανταγωνισμού. Και θα συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μεριμνήσουμε για τη διαφύλαξη του κοινοτικού χαρακτήρα της κοινή γεωργικής πολιτικής. Και μερικά σχόλια ακόμη. Ο εισηγητής είπε ότι θα καταθέσει τροπολογία για την περιφερειακή ανάπτυξη και το βαθμό απορρόφησης των κονδύλιων. Εκτός και αν δεν σας κατάλαβα καλά. Γιατί για την αγροτική ανάπτυξη υπάρχει μεγάλος βαθμός απορρόφησης. Και το αναγνωρίζει και η έκθεση ότι δεν είναι πρόβλημα απορρόφησης ε, της αγροτικής ανάπτυξης, αλλά ρυθμού δαπανών και συμφωνούμε ότι η ψηφιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες που μπορούν να βοηθήσουν και για την ελάφρυση του διοικητικού άχθους αλλά και για την οικολογικοποίηση της ΚΑΠ είναι ευπρόσδεκτες και συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη στο σημείο αυτό. Σε ό,τι αφορά την κατανομή των άμεσων ενισχύσεων και αυτό το καλύπτουμε στην, στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, ήθελα να πω ότι αναγνωρίζω ότι στη δική σας πρόταση μιλάτε για την ανείχνευση και την αποτροπή της απάτης και έμφαση στο κράτος δικαίου, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την υφαρπαγή γεών. Ε, έχουμε δηλώσει ότι όταν μιλούμε για υφαρ, υφαρπαγή γεών και ο κύριος Δόρφων αναφέρθηκε στο άρθρο των, ε, Financial Times, θα πρέπει να δούμε αν πρόκειται όντω για απάτη. Και όσο αφορά τα συστήματα διαχείριση και ελέγχου των κρατών μελών, αυτό ουσιαστικά κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακολουθεί στενά κατά πόσο ακολουθούνται οι κανόνε στα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ζητήματα του κράτου δικαίου, υπάρχουν και πάλι νομοθετικέ διατάξει που διέπουν την κυριότητα των γεών ή την δυνατότητα αγορά γεών στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι θέμα κράτους δικαίου και έχουμε και σχετική πρόταση για την ΚΑΠ μετά το 2020. Και επαγρυπνούμε και σε θέματα κράτους δικαίου. Και μάλιστα ότι καταγγελίες υπάρχουν ή πληροφορίες ε, δεν ε, περνάνε στον τούκου, τις διερευνούμε εις βάθος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν ο εισηγητή θέλει να ξαναλάβει το λόγο. Από ό,τι βλέπω όχι. Ω εκ τούτου, επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι η 6η Δεκεμβρίου στη 1 η ώρα το μεσημέρι είναι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των τροπολογιών και θα εγκρίνουμε την έκθεση στι 23 Ιανουαρίου. Ε, η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή οφείλει να υιοθετήσει την ε, έκθεση μέχρι τι 20 Φεβρουαρίου. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα της μερίσιας διάταξης που είναι η πολιτική ανταγωνισμού. Και επ' αυτού έχουμε την ετήσια έκθεση του 2019. Ως ε, Επιτροπή Γεωργίας από το 2016 έχουμε υιοθετήσει μια παράδοση, δηλαδή να συντάσουμε γνωμοδότηση η συγγήτρια κυρία Καβαλιές, είναι η συγγήτρια και έχει συντάξει σχέδιο έκθεσης το οποίο και επιθυμεί να μας παρουσιάσει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να υπενθυμίσω ότι η πολιτική ανταγωνισμού θα πρέπει να επιτρέψει την υλοποίηση των στόχων της κοινής πολιτικής εφαρμόζοντας φυσικά την υπεροχή της αγροτικής πολιτικής ε, έναντι των κανόνων του ανταγωνισμού, όπως ε, επιβεβαιώνει η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόσφατα και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, κάτι που άλλωστε δικαιολογείται από τις ιδιαιτερότητες της γεωργίας. Είναι σημαντικό να μεριμνήσουμε ώστε η πολιτική ανταγωνισμού συμβάλλει όντως την ενίσχυση του θέση, της θέσης του Γεωργού εξασφαλίζοντας δίκαια αποτελέσματα και για τους καταναλωτές αλλά και για τους παραγωγούς. Ε, με βάση αυτές τις αρχές κατά νου, συνέθεσα την γνωμοδότησή μου ε, και θα ήθελα να σας πω ότι λόγω των, κανόνων ήταν περιορισμένη. Θα πρέπει λοιπόν να τη συμπληρώσουμε και να προσέξουμε όχι μόνο το θέμα της Πολιτική ανταγωνισμού και τη πολιτική γεωργίας, αλλά και κάποια άλλα σημεία που κατά τη γνώμη μου χρήζουν επισήμασης. Επίσης, ε, όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση ε, ε, για, την ετήσια έκθεση ανταγωνισμού, θα μιλήσω για τις κρατικές ενισχύσεις για τη στήριξη και εγκατάσταση της ευρυζωνικότητας. Οι κρατικές αυτές ενισχύσεις είναι πολύ σημαντικές λόγω της μεγάλη σημασία που έχει η καινοτομία και η ψηφιοποίηση στη γεωργία και που θα χρειαστούν για να μην μείνουν πίσω οι αγροτικές ζώνες. Και γι' αυτό θα καταθέσω κάποιες τροπολογίες και καλώ τους συναδέλφους να κάνουν το ίδιο. Πάντως, εγώ τόνισα κάποια σημεία στη γνωμοδότησή μου που κατά τη γνώμη μου είναι τα πιο σημαντικά για τον τομέα της γεωργίας στα πλαίσια και της πολιτικής ανταγωνισμού και της ανταγωνιστικότητας. Ένα από τα βασικά σημεία αφορά τις οργανώσεις παραγωγών και τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών. Και θα ήθελα επ' ευκαιρία να χαιρετήσω την έκθεση, τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επικεντρώθηκε στους τομείς των αρτρέων καλλιεργειών, του βοήου κρέατος και του ελαιολάδου με βάση έρευνες που έγιναν στον κλάδο και που επιβεβαιώνουν τη σημασία που έχουν οι οργανώσεις αυτές στην ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού σε τρόφιμα και στην προάσπιση ενός δίκαιου βιωτικού επίπεδου για το γεωρικό πληθυσμό. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω, αλλά θα ήθελα παρόλα αυτά να εξάρω την ε, υιοθέτηση την έγκριση τη οδηγία για την καταπολέμηση των αθέμητων εμπορικών πρακτικών είναι πολύ σημαντικό για να εξασφαλίσουμε καλύτερη ισορροπία στην διαπραγματευτική ισχύ και των γεωργών. Βέβαια, η μεταφορά τη οδηγία αυτή στην ένωμη τάξη εναπόκειται στα κράτη-μέλη. Είναι σημαντικό όμω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθήσει αυτή τη διαδικασία και να προωθήσει ε, την αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών και την ανταλλαγή απόψεων για αυτέ. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε την ισορροπία μεταξύ των διαφόρων κρίκων τη αλυσίδα εφοδιασμού για να μην θέσουμε σε κίνδυνο ορισμένους κρίκους της Θα πρέπει λοιπόν να αναλύσουμε τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να έχουν οι συμμαχίες των αγοραστών σε ό,τι αφορά τη διατάραξη αυτής της ισορροπίας, γιατί ήδη έχουμε ε, σημαντικές ενδείξεις για τη διατάραξη αυτή τη ισορροπία και τι αρνητικέ συνέπειε, ε, όπω δείχνουν κάποιε έρευνε που έχουν ξεκινήσει από τι αρχέ ανταγωνισμού. Είναι σημαντικό λοιπόν επ' ευκαιρία και χαιρετίζω το σεμινάριο που οργάνωσε για το θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα. Επίσης, ε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να προτείνουμε την ε, ε, οργανική αλλαγή που πρότεινε, στο, την αλλαγή στο οργανόγραμμα που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, το θέμα της μεταφοράς των θεμάτων κάποιων γεωργικών και δασοκομικών από την Επιτροπή Γεωργίας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλα αυτά τα θέματα στην ε, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, γιατί αυτή η Γενική Διεύθυνση έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να ε, επεξεργαστεί και να παρακολουθήσει τις, ε, την εξέλιξη των σημαντικών και ιδιαίτερων αναγκών που έχει ο κλάδος. Αυτά και περιμένω τις τροπολογίες σας για να τις συμπεριλάβω στην γνωμοδότησή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς ε, πάρα πολύ για την παρουσίαση του σχεδίου της έκθεσης ε, και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον ε, σκιώδη συγκτή του ΕΛΚ, τον συνάδελφο κύριο Μπούντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εισήγησή της <clears throat> και επίσης και για τη μελέτη σχετικά με τις οργανώσεις παραγωγών. Διαπιστώνουμε ότι το επίπεδο της οργάνωσης ποικίλει από τη μία χώρα στην άλλη. Η μελέτη επισημαίνει ότι το βασικό αίτιο για τη δημιουργία αυτών των οργανώσεων παραγωγών, ο βασικός λόγος είναι για να <clears throat> διασφαλίσουμε την πρόσβαση σε κάποιες αγορές και να διασφαλίσουμε και τη δική τους την ύπαρξη. Σε συζητήσεις που είχα με γεωργούς από τη Ρουμανία, το Βέλγιο και άλλες χώρες, πραγματικά εντυπωσιάστηκα από το ότι ανέφεραν το θέμα των τιμών. Τα τελευταία 20 χρόνια εξακολουθούν να έχουν την ίδια τιμή γάλακτος παρότι οι τιμές, οι εμπορικές τιμές είναι πολύ ψηλότερες. Νομίζω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι γεωργοί αλλά και οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να είναι εκείνοι που να στιγματιστούν ως οι άμεσα εποφελούμενοι από τις υψηλότερες τιμές για να διαφυλαχθούν οι πολιτικές ανταγωνισμού, θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στους ε, γεωργούς ε, αλλά και γενικότερα να περιστούν οι ανισορροπείς ανάμεσα στους άμεσα ενδιαφερόμενους και να συσταθούν ίσες ευκαιρίες ανταγωνισμού στο μέλλον θα πρέπει να έχουμε διαφορετική προσέγγιση στο θέμα των τιμών, ε, να έχουμε τιμές ε, που να είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στην αγορά, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική καινοτομία και τις ε, επιπτώσεις στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω και το συσχετισμό ανάμεσα στην τιμή παραγωγής και την τελική τιμή πώλησης, διότι δυστυχώς ε, προκύπτει μια κατάσταση όπου οι γεωργοί πολλούν τελικά σε τιμή που είναι και κάτω από την ε, τιμή παραγωγής. Επόμενη η συνάδελφος ε, Αλίε Βαβέλη. Κύριε Πρόεδρε, το σχέδιο έκθεσης ε, είναι μια πολύ καλή βάση για τη δουλειά μας. Περιλαμβάνει πολλά και σημαντικά θέματα και θα θέλαμε και εμείς βέβαια από πλευράς μας ε, να προσθέσουμε κάποια θέματα γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να ελέγχουμε τα φυτικά φάρμακα, τα ζυζανιοκτώνα. Εξάλλου, υπογραμμίζουμε το ότι είναι απαραίτητο να ε, θεσπιστεί έγκαιρα μεταβατική νομοθεσία έτσι ώστε να αποφύγουμε την ένταση στις ε, αγορές. Και ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι η στρατηγική που λέει απευθείας από την παραγωγή, από το γεωργό στην κατανάλωση. από την ε, γεωργική εκμετάλλευση κατευθείαν στο πυρούνι σε εισαγωγικά. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια νέα στρατηγική σχετικά με τις οργανώσεις αγοράς. Και επόμενος ε, από το ECR, παρακαλώ, έχετε το λόγο ο κύριος Ρούισεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτό το πολύ καλό σχέδιο γνωμοδότησης ε, είναι πολύ καλό το σχέδιο αυτό. Αναφέρονται τα σημαντικότερα θέματα που έχουν σχέση με τον ανταγωνισμό. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε τη θέση του Γεωργού στην αλυσίδα εφοδιασμού. Και είναι πολύ σωστό το ότι η συγγήτρια επισημαίνει τον ιδιαίτερο ρόλο της Γεωργίας γιατί είναι απαραίτητο να υπάρξουν απλουστεύσεις ε, έτσι ώστε να ενισχυθεί η παραγωγή και να ενισχυθεί και η ε, αλυσίδα εφοδιασμού με τελικό στόχο να επιτευχθούν καλύτερες τιμές. Αυτό που μου αρέσει καλύτερα στην γνωμοδότηση είναι ότι επισημαίνονται διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν σχέση με τη βιωσιμότητα. Είναι σημαντικό και στο θέμα αυτό να επενδύσουμε έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στους γεωργούς να συνάψουν συμφωνίες σχετικά με τη βιωσιμότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ωφελήσει την κοινωνία ευρύτερα, τους καταναλωτές ειδικότερα και νομίζω ότι είναι σημαντικό να προβλέψουμε τέτοιες πρωτοβουλίες βιωσιμότητας και να προβλέψουμε και ε, εξαιρέσεις ε, από τις διατάξεις περί ανταγωνισμού. Σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεση. Πρόεδρος, οι υπόλοιπε πολιτικές ομάδες ε, δεν έχουν προτείνει σε εισηγητέ. Δεν ξέρω, θέλει κάποιος να λάβει το λόγο εκ μέρου της πολιτικής ομάδας. Αν όχι, έχουν ζητήσει τρεις ακόμα το λόγο. ένα εξ αυτών, ο συνάδελφος Ρουπέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγητριά μας γιατί είναι πολύ αξιόλογο το, θε... το πόνημά της και το θέμα είναι πολύ σημαντικό και όχι μόνο για τους παραγωγούς αλλά και για τους καταναλωτές. Έχουμε μεγάλο αριθμό κατοίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω από 500 εκατομμύρια. Επίσης, ε, οι εμπορικέ μας συναλλαγές και το ενδοκινοτικό εμπόριο, αλλά και οι εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια ανταγωνιστικότητα της γεωργίας μας ε, και εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα θέματα ανταγωνισμού και γεωργίας είναι άρρηκτα ε, δεμένα μεταξύ τους. Και φυσικά χρειάζεται απαραίτητος προϋπολογισμός και για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας στη Γεωργία. δεν ΔΕΜΗ δεν πρόκειται να λύσουμε τα προβλήματά της. Ας μην ξεχνούμε ότι οι Γεωργοί με πολύ ιδιαίτερες συνθήκες καλούνται να ανταγωνιστούν τους ε, υπόλοιπους Γεωργούς. Και το θέμα των τιμών και του προσδιορισμού των τιμών είναι πολύ σημαντικό, γιατί η τιμή είναι τα δύο τρίτα περίπου του εισοδήματο του Γεωργού. Και δεύτερο ζήτημα είναι το ζήτημα των ενισχύσεων. Θα πρέπει να έχουμε σωστέ ρυθμίσει για τι ενισχύσει, ώστε να εξασφαλιστούν συνθήκε ε, ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών. Γιατί αν είναι διαφορετικά τα επίπεδα των, ε, κρατικών, των εθνικών ενισχύσεων για του γεωργούς, διαταράσσεται ο θεμητό ανταγωνισμό. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει δίκαιο και θεμητό ανταγωνισμό μεταξύ των γεωργών. Αυτό με ενδιαφέρει κατάλληλες συνθήκες για όλους τους γεωργούς στον ανταγωνισμό. Και θέλουμε αυτές οι συνθήκες ε, ισότιμου ανταγωνισμού να αναφέρονται στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά το 2020. Πριν από λίγες εβδομάδες, χιλιάδες Λιθουανοί ε, Γεωργοί κατέκλυσαν τους δρόμους της Λιθουανίας με τα τρακτέρ τους και διαδήλωσαν. Βλέπετε εδώ τις φωτογραφίες. Ε, ε, οι Γεωργοί διαμαρτύρονται γιατί θεωρούν ότι υφίστανται αθέμητο ανταγωνισμό. Επίσης το επίπεδο άμεσων ενισχύσεων στις χώρες Βαλτικής είναι το χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι Λιθουανοί κτηνοτρόφοι σήμερα παράγουν μόνο ε, τις μισές ποσότητες ε, ε, που χρειάζονται για την ε, εσωτερική κατανάλωση. Και έτσι οι Λιθουανοί καταναλωτές ε, αναγκάζονται να αγοράσουν εισαγόμενα προϊόντα. Επίσης, η τιμή του γάλακτος έχει καταποντιστεί. Η θέση των Λιθουανών γεωργών και κτηνοτρόφων είναι ότι υφίστανται αθέμητο ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι που δεν ισχύει για όλους τους γεωργούς. Οπότε θα πρέπει να βρούμε λύσεις που όχι μόνο θα διασφαλίζουν αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο στους ε, εν ενεργεία αλλά θα προσελκύσουμε με τις ευνοϊκές αυτές συνθήκες και νέους γεωργούς στο κλάδο. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου όχι μόνο βράχη και μέσο πρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα τη γεωργία. Καλή η γνωμοδότηση, θα καταθέσουμε και εμείς τροπολογίες. Ευχαριστώ κύριε Ροπέ. κύριε Αγγιλέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τη συνάδελφο Ισαβέλ Καραβαλιάης γιατί η έκθεση της ε, είναι πολύ αξιόλογη και αποτελεί μια καταπληκτική ε, αφετηρία για τη συζήτηση της πολιτικής ανταγωνισμού στη Γεωργία. Και είναι από τις ε, σημαντικότερες συζητήσεις που έχουμε μπροστά μας. Θα πρέπει λοιπόν να αφιερώσουμε πολύ χρόνο για να συζητήσουμε ένα από τα πιο φλέγοντα προβλήματα της γεωργίας, που είναι οι χαμηλές τιμές παραγωγού, οι χαμηλές τιμές δηλαδή που λαμβάνουν οι γεωργοί στην τροφική αλυσίδα. Και χαίρομαι που έχουμε επιτέλους την οδηγία για την καταπολέμηση των αθέμητων εμπορικών που δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί από όλα τα κράτη-μέλη, αλλά βλέπουμε πώς εδώ και χρόνια γεωργοί και κτηνοτρόφοι λαμβάνουν ε, τιμές για τα προϊόντα τους που είναι αυτές που είχαν πριν από 10-20 χρόνια. Είναι αδύνατο και απαράδεκτο αυτό. Θα πρέπει λοιπόν ε, να συζητηθούν και να εξεταστούν αυτά τα θέματα όχι μόνο στη δική μας Επιτροπή, αλλά και πέραν αυτής. Οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι μας καλούνται να εφαρμόσουν πολύ υψηλέ προδιαγραφές και πρότυπα, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και είμαστε υπερήφανοι για τι υψηλέ μα προδιαγραφές, αλλά όλες αυτές οι απαιτήσει φέρνουν τη γεωργία και κτηνοτροφία σε μια δυσβάσταχτη κατάσταση και φαίνεται ότι αγνοούμε το πρόβλημα των πολύ χαμηλών τιμών. Ενώ οι καταναλωτές φυσικά ε, και η ε, Επιτροπή χαίρεται που έχουμε χαμηλέ τιμέ ε, για τον καταναλωτή γιατί σκέφτεται και τα δικά του συμφέροντα. Το θέμα είναι ότι οι καταναλωτές δεν αποφελούνται από αυτές τις χαμηλές τιμές παραγωγού, γιατί ναι μεν πλήττονται οι γεωργοί από τις χαμηλές τιμές που λαμβάνουν για τα προϊόντα τους, αλλά οι καταναλωτές εξακολουθούν να ε, πληρώνουν υψηλέ τιμές για να αγοράζουν τα τρόφιμά τους. Δεν συμφωνούμε με την πολιτική αυτή και νομίζω ότι είναι πολύ κακό μήνυμα οι εθνικές οι κρατικές ενισχύσεις στη Γεωργία και τη δασοκομεία να περάσουν από την Γενική Διεύθυνση Γεωργία στη Γενική Διάθεση Ανταγωνισμού. Όχι, είναι πολύ κακό το μήνυμα. Θα πρέπει να παραμείνουν στην Επιτροπή, στην Γενική Διάθεση Γεωργία. Δεν μπορούμε τι εθνικέ ενισχύσει, κρατικέ ενισχύσει για τη Γεωργία να τι μεταφέρουμε στην πολιτική ανταγωνισμού, στην Γενική Διάθεση Ανταγωνισμού. Γιατί θα δώσουμε το μήνυμα που έχουν ήδη λάβει οι Γεωργοί ότι τι μεταφέρετε στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και θέλετε να τι περιορίσετε ή να τι καταργήσετε. Όχι. Δεν θα πρέπει να περικόψουμε τι κρατικέ ενισχύσει στη Γεωργία και νομίζω ότι ε, προς τα εκεί βαδίζουμε αν μεταφέρουμε αυτές τις αρμοδιότητες στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας που ήταν προηγουμένως. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα και φυσικά μέσω της έκθεσής μας ε, να στείλουμε και εμείς ένα χειρό μήνυμα ότι δεν θα πρέπει κρατικέ ενισχύσει για την Γεωργία να περάσουν στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, γιατί η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού είναι κατά των κρατικών ενισχύσεων και άρα θα τι περικόψει δραστικά ή θα τι καταργήσει. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εμεί βρισκόμαστε εδώ για να λύσουμε τα προβλήματα των γεωργών. Και γι' αυτό θα πρέπει να εξισορροπηθούν οι καταστάσεις μεταξύ των διαφόρων κρίκων της τροφικής αλυσίδας. Και Συμφωνώ και με την πρόταση για τις οργανώσεις παραγωγών. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμω με τι οργανώσεις παραγωγών οποροκυπευτικών. Οι ελάχιστε προϋποθέσεις κάποιων χωρών για τη διαπίστευση οργανώσεων παραγωγών επιτρέπουν ε, κάποια δυσανάλογα συστήματα. Δεν μπορούμε να μειώνουμε τις εθνικές, ε, τις εθνικές ε, για τις οργανώσεις παραγωγών που ουσιαστικά αλλοιώνουν την κατάσταση και πλήττουν τους γεωργούς και όχι τους διανομής και τους πελάτες τους. Προσοχή! Με τις απαιτήσει αυτές που είναι εθνικές απαιτήσει, πολλές φορές αλλοιώνουμε τη λειτουργικότητα και τη χρηστικότητα του σημαντικού μέτρου που είναι οργανώσει των παραγωγών και που χρειάζονται. Θα πρέπει λοιπόν να τους αποδυναμώνουμε. Στην Ισπανία έχουμε σημειώσει αρκετή πρόοδο, αλλά θα πρέπει οι απαιτήσει στο μέλλον να είναι υψηλέ. Γιατί πρόκειται για μια οργανωτική ε, δομή που χρειάζεται υπέρ των ε, παραγωγών, των γεωργών, όχι υπέρ των εμπόρων, των διανομέων και των πελατών τους. Γι' αυτό αναγνωρίζουμε τις οργανώσεις παραγωγών και για κανένα άλλο λόγο. Προσοχή λοιπόν με το επίπεδο των απαιτήσεων. Ελπίζω να γίνει κάποια έκθεση για να δούμε πώς στο μέλλον μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το σωστό εργαλείο που είναι η οργανώση παραγωγών. Αλλά προσοχή με τα εθνικά κριτήρια και τις απαιτήσει. γιατί θα ακολουθήσουμε λάθος δρόμο αν έχουμε τα ίδια πράγματα όπως και με τα κριτήρια για τα εθνικά. Ευχαριστώ αγαπητή συνάδελφα. Συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά του του Είναι πολύ επίκαιρη αυτή η γνωμοδότηση και θα πρέπει να συμπεριλάβουμε ε, αναφορές ε, για τις στρατηγικές και να προσπαθήσουμε να ε, έχουμε μια αναφορά για τον ανταγωνισμό σε θέματα προτύπων στις τρίτες χώρες. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό θέμα για τους γεωργούς. Ειδικά όταν κάνουμε αναφορά για τα βιώσιμότητα στα τρόφιμα. Ε, από τη φάρμα κατευθείαν στο πυρούνι, στρατηγική αυτή, γιατί ο... η στρατηγική του δεν θέτει ένα τίμημα στα δημόσια αγαθά επίσης, να συμπεριλάβουμε και την κλιματική διάσταση, οι αγρότες, διαμαρτύρονται οι αγρότες στην Ιρλανδία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία και σε άλλες χώρες. Είναι ανήσυχοι οι γεωργοί σχετικά με αυτά που συμβαίνουν. Θεωρούν ότι θα πρέπει να κάνουν περισσότερα για το περιβάλλον, όμως ο προπολογισμό έχει μειωθεί από την ε, κοινή γεωργική πολιτική και επίσης η αγορά δεν πληρώνει για την ε, παράδοση αυτών με την ευκαιρία αυτής της γνωμοδότηση θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτά τα θέματα και η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού δεν είναι φιλικά προσχήμενη στους γεωργούς γιατί είναι πολύ στενή η έννοια του ανταγωνισμού όπως την αντιλαμβάνονται δεν λαμβάνουν υπόψη τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τη γεωργία, με την ε, φύση, άρα θα ε, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη αναγνώριση για το φαγητό, που είναι ένα θεμελιώδες αγαθό για την ε, επιβίωση και το τρέχον μοντέλο που υποχρεώνει τους αγρότες να παράγουν περισσότερα για λιγότερα είναι κάτι μη βιώσιμο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, συνάδελφος Δεκάστρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τους προηγούμενους συντέλφους ότι η συνάδελφος Ισαμπέλα έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Ε, το θέμα ε, τέθη από την προλήσα την κυρία Αγγιλέρα και θα ήθελα και εγώ να το ξαναεπαναφέρω. Δηλαδή ε, είναι απαραίτητο να τοποθετηθούμε στο θέμα των κρατικών ενισχύσεων. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτή η γνωμοδότηση μπορεί να συμπεριλάβει αυτό το θέμα, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν κάποια νομοθετική φύσεως θέματα σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, να συνδεθεί με το άρθρο 42 της συνθήκης, για να μπορούμε να έχουμε μια μεγαλύτερη ευελιξία, η οποία θα μπορούσε να χορηγηθεί στα κράτη-μέλη, αλλά να διασφαλιστεί αυτό το εργαλείο. Κατά τα άλλα, τα είπε η Στάσπος κυρία σε πράγματι έχουμε την οδηγία ε, κατά των παράνομων εμπορικών ε, πράξεων. Έχουμε επίσης ε, το θέμα του ανταγωνισμού στη Γεωργία. Όλα αυτά είναι πολύ ουσιαστικά. Ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το ανέφερε η Άσπρο Ιζαμπέλ, Βέβαια, προσπάθησε να διευκρινίσει ότι οι διατάξεις συνδέονται με, την, με τις ιδρυτικές συνθήκες, άρα δηλαδή δεν υπάρχει κανένας είδους ε, κατάχρηση από πλευράς οργανώσεων των παραγωγών ή των ενδιάμεσων οργανώσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή, στον κύριο Σόφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα αναφερθώ σε κάποια θέματα που θύχτηκαν. Να υπογραμμίσω τη σημασία του θέματος των τιμών που πολλά μέλη εδώ έθιξαν και την θέση των γεωργών στην αλυσίδα. Είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή συγκεκριμένα ε, είναι κάτι πάνω στο οποίο έχουμε εργαστεί τα τελευταία δέκα χρόνια και υπάρχει μία έκθεση από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού που αναλύει τι πράττουν οι γεωργοί σε αυτό το θέμα και η λύση μακροπρόθεσμα είναι στι οργανώσει παραγωγών. Οι κανονισμοί μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, αλλά η πραγματική απάντηση, όπω λένε αυτοί, δεν είναι εμείς όπως λένε οι αγρότες, αλλά οι οργανώσεις παραγωγού που θα βελτιώσουν τη θέση τους παρέχοντας τους υπηρεσίες όπως ε, τη διανομή, ε, ποιοτικού ελέγχους που θα τους δώσουν διαπραγματευτική δύναμη σε σχέση με τους αγορευτές και που θα μειώσει το κόστος, γιατί η απάντηση δεν ε, έχει να κάνει μονάχα με τις τιμές αλλά και με το κόστος γιατί ε, τα έσοδα τους είναι τιμές μείων κόστος, όχι μόνο τιμές. Αυτό μας δείχνει λοιπόν το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε ε, από την πλευρά των γεωργών και πιστεύουμε περισσότεροι γεωργοί να συμμετέχουν σε αυτή την εξέλιξη και η Επιτροπή το υποστηρίζει αυτό το σχέδιο και έχει ταχθεί υπέρ των νέων μεταρρυθμίσεων στα εθνικά προγράμματα, ώστε να έχουν τη στήριξη ε, οι αγρότες, να έχουν τους κατάλληλους κατάλληλες οργανώσεις ε, που θα τους βοηθήσουν όσα ε, τη μεταφορά των αρμοδιότητων από την ε, Γενική Διεύθυνση Άγκρη στην Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Οι αποφάσεις αυτές έχουν να κάνουν με τις αποφάσεις του Κολεγίου των Επιτρόπων. Πρώτον, η νομοθεσία δεν θα αλλάξει, παραμένει ως έχει. Η νομική βάση είναι επίσης η ίδια, οι κανόνες είναι οι ίδιοι και μπορούν να αποφασιστούν οι κανόνες από την ε, συνέλευση αυτή που χρειάζεται. Δεν υπάρχουν αλλαγές στους κανόνες όμως, όπως είπαμε. Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού έχει συμμετάσχει ήδη στην ε, εφαρμογή ε, κανόνων σχετικά με τα αγροτικά, αγροτικών προϊόντων και έχουν συνεργαστεί επίσης οι δύο γενικέ διευθύνσεις, η ε, Άγκρη με την ε, Γενική Διευθύνση Ανταγωνισμού και να είστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουν ε, να συνεργάζονται και ότι θα υπάρχει μια συνέχεια όσον αφορά τι κρατικές ενισχύσει. και μια σταθερότητα. Σε σχέση με τις, πληρωμέ, με τις ενισχύσεις, και του γεωργού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε στην επόμενη μεταρρύθμιση τη ε, ΚΑΠ. Θα επανέλθουμε λοιπόν σε αυτό το θέμα. Υπήρξαν κάποια σχόλια για, τη βιωσιμ... για, τις πρωτοβουλίες βιωσιμότητας. Είναι πολύ σημαντικό και αντίθετα με αυτά που έχουν υποθεί οι, οι υπηρεσίες ανταγωνισμού τα στηρίζουν αυτά τα προγράμματα. Ε, έχουμε το παράδειγμα του Chicken of Tomorrow στην Ολλανδία. Ε, στην περίπτωση αυτή βοηθάνε τους ε, γεωργούς Μπορεί να μην υπάρχει βελτίωση στις τιμές, όμως ε, το σύστημα αλλάζει με διάφορες πρωτοβουλίες και κατάφεραν να πετύχουν βελτιώσεις στο θέμα της βιωσιμότητας όμως τιμέ ήταν υψηλέ για αυτού που ήταν πρόθυμοι να εφαρμόσουν αυτές τις αλλαγέ. Η Γενική Διευθυνσία Ανταγωνισμού και η Επιτροπή δεν εμποδίζουν αυτές τις διαπραγματεύσεις, αλλά βοηθούν τους αγρότες για την ε, αύξηση των εσόδων τους. Όσον αφορά την οριζόντια συνεργασία, υπάρχει ένα σαφές ε, πλαίσιο και κατευθυντήριε γραμμές. αυτέ οι κατευθυντήριε γραμμές είναι υπό αναθεώρηση. Μέχρι τον Φεβρουάριο του επόμενου έτου, υπάρχει μια δημόσια διαβούλευση στην οποία μπορεί να απαντήσει ο κάθε ε, ενδιαφερόμενος και θα υπάρξει μια πλήρη αναθεώρηση αυτών των ε, κατευθυντήριων γραμμών μέσα στο επόμενο διάστημα, διάστημα οπότε είναι κατάλληλη στιγμή για να, προτείνετε, ε, να κάνετε προτάσεις, να υποβάλλετε προτάσεις για τον σχεδιασμό των ε, κανόνων για, την, ε, για τον οριζόντια συνεργασία όσον αφορά τη βιωσιμότητα και άλλα θέματα. Και με αυτά νομίζω ότι απάντησα σε όλα τα θέματα που θύχτηκαν. Αν υπάρχει κάποια άλλη ε, ερώτηση, είμαι πρόθυμος να απαντήσω. Ευχαριστώ την Επιτροπή. Θα δώσω και πάλι το λόγο στην εισηγήτρια. Θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους, για τις παρατηρήσεις τους. Φυσικά υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης και εμπλουτισμού της γνωμοδότησης. Και περιμένω τις τροπολογίες σας για να τις συμπεριλάβω στη γνωμοδότησή μου. Και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα δικά της σχόλια. Δεν έχω τίποτα άλλο κύριε Πρόεδρε να προσθέσω. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Απλά να επισημάνω ότι η καταληκτική ημερομηνία για κατάσταση απολογιών είναι 10 ε, Δεκεμβρίου, μία ώρα το μεσημέρι. Όπω είπα, τον Ιανουάριο θα γίνει δεκτή η ε, έκθεση και στις 18 Φεβρουαρίου η Καθήλυνα Αρμόδια Επιτροπή ε, θα πρέπει και εκείνη να υιοθετήσει την έκθεση. Πάμε λοιπόν στο σημείο υπαριθμών 5 της ημερήσιας διάταξης που είναι ο καθορισμός, η θέσπιση του προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων και τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Ήδη λοιπόν από τον τίτλο βλέπετε ότι το θέμα δεν είναι και τόσο απλό. Η συγγήτρια είναι η κυρία Σμιτμπάουα και τώρα βρισκόμαστε ε, το ότι έχουμε ολοκληρώσει τον δεύτερο τριμερή διάλογο. Καθήλυνα αρμόδια επιτροπή είναι αυτή της ε, κοινή αγοράς. Εμείς ε, συμμετέχουμε βέβαια με βάση το άρθρο 57 και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην άρθρο κυρία Σμιτ Μπάουα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως ε, αναφέρατε, ο δεύτερος τριμερής ε, διάλογος έλαβε χώρα στις 18 Νοεμβρίου. Κάναμε κάποια πρόοδο, περιορισμένη βέβαια. Ε, ο κατάλογος των θεμάτων επί των οποίων συμφωνήσαμε, ο κατάλογο αυτό εγκρίθηκε. Υπάρχουν κάποια πολιτικής φύσεως θέματα και εμείς ως Επιτροπή Γεωργίας είμαστε αρμόδιοι. Αυτά συζητήθηκαν τρία άρθρα. Δηλαδή, το ένα είναι ο τομέας, το πεδίο εφαρμογή, ο δεύτερο τομέα είναι τι διατάξει περί συγχρηματοδότηση. και το τρίτο θέμα που συζητήθηκε είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο. Το άρθρο για το πεδίο εφαρμογή, ε, εκεί οι απόψει ε, του συνομοθέτη είναι πολύ περιορισμένε. Ε, έπρεπε να κάνουμε κάποιε εκ των προτέρων, να συμφωνήσουμε σε κάποια θέματα για να μπορούμε να επιτύχουμε το τελικό μα αποτέλεσμα. Και τώρα σε τεχνικό επίπεδο αναθέσαμε να εξετάσουν το πώς ακριβώς μπορούν να συνδυαστούν οι προτάσεις όλων των θεσμών. Όσον αφορά στο άρθρο για τις διατάξεις συγχρηματοδότησης για θέματα φυτοϊγιεινής, το Συμβούλιο προσπαθεί να αντιστρέψει την αρχή της χρηματοδότησης. Δηλαδή επιθυμεί να, έχει, να ορίσει κατώτατα όρια χρηματοδότησης, όμως η Επιτροπή διαφωνεί κάθετα, γιατί αυτό θα μπορούσε να αποτελεί ε, το να, θέσει, να τεθεί σε κίνδυνο ο προϋπολογισμός. Βεβαίως, το Συμβούλιο πιστεύει ότι με εφαρμοστική πράξη μπορούν να αλλάξουν ε, τα, οι συντελεστές χρηματοδότησης. Το ε, Κοινοβούλιο διαφώνησε κάθετα. Εξάλλου, ε, δεν θα πρέπει όλα αυτά να είναι δυνατά μέσω ενός εφαρμοστικού κανονισμού. Το, Συμβούλιο, με συγχωρείτε, το Κοινοβούλιο επισήμανε ότι αυτό το τόσο σημαντικό θέμα πρέπει να συζητηθεί σε πολιτικό επίπεδο. Και το τελευταίο θέμα, το οποίο αφορά τις αρμοδιότητες μας ως Επιτροπή, έχει σχέση με το πλαίσιο χρηματοδότησης για το πρόγραμμα της κοινή αγοράς. Ήδη κατά την πρώτη συνεδρίαση διεφάνει ότι το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή δεν θέλει να συζητήσει για αριθμούς ε, του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου διότι θεωρεί ότι ε, υπάρχουν αρκετές ελλείψεις στον προϋπολογισμό και γι' αυτό το λόγο συμφωνήσαμε ότι τελικά στις διαπραγματεύσεις δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο πρόοδου αν δεν συζητηθεί ο προϋπολογισμός. Και γι' αυτό το λόγο οι διαπραγματεύσεις ε, πάγωσαν ε, επαόριστον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την συνάδελφο κυρία Σμιτ Πάουα. Δεν ξέρω αν κάποιος επιθυμεί να λάβει το λόγο επ' αυτόν που ακούσαμε. Από ό,τι βλέπω όχι. παρότι τα νέα δεν ήταν και ιδιαίτερα ευχάριστα, τι να κάνουμε. Αλλά εντάξει, κλείνουμε και αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης και ως εκ τούτου διακόπτεται τώρα η επίσημη συνεδρίαση μέχρι σήμερα το απόγευμα ε, στις 2.30 όπου θα συνεχιστεί η δημόσια συνεδρίαση από τις 15.30 έχουμε την ακρόαση για την ΚΑΠ η συνεδρίαση των συντονιστών θα λάβει χώρα από τις 10.30, αλλά ο συνήθως θα είναι και κλεισμένων των θυρών. Σας ευχαριστώ πολύ.